get Hello everybody. Ας αρχίσουμε. Καλημέρα σε όλους και καλώς ορίσατε. Και πάλι. We have to finish the... Έχουμε κάτι θεματάκι ακόμα για σήμερα. Το πρώτο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το σχέδιο ψηφίσματος για την ε, ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα άτομα με αναπηρίες μετά το 2020. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια. Η σημερινή στρατηγική, όπως όλοι γνωρίζετε, φέτος λίγη και έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές ε, είναι τεράστιες οι διαφορές σύμφωνα με την έκθεση εφαρμογής ε, από κράτος σε κράτος. Πώς φέρεται και πώς φροντίζει ε, τα αμαία κάθε χώρα. Θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα εξωφρενικό επισέδιο στην Τσεχία. Οχτώ άτομα με πνευματική αναπηρία έχασαν τη ζωή τους σε μια πυρκαγιά. Η ε, συνήγορος του πολίτη στη Τσεχία επανειλημμένα ε, έχει ε, ειδοποιήσει ε, ότι υπάρχει πρόβλημα στα ιδρύματα στη Τσεχία ε, για ανθρώπους με πνευματική αναπηρία, για λόγους ασφαλείας. Και οχτώ έχασαν τη ζωή τους σε μια πυρκαγιά, είπαμε. Τα τσεχικά ιδρύματα δεν προσφέρονται για μακροχρόνια διαβίωση και είναι κίνδυνο στα ίδια τα ιδρύματα για τη ζωή των τροφίμων η αποϊδρυματοποίηση δεν μπορεί να είναι κάτι που θα το γράφουμε σε χαρτιά. Δεν μπορεί κάποιοι ε, άνθρωποι να είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν σε ένα ίδρυμα 50 άτομα με πνευματική αναπηρία. Και ε, περίπου 50 και πλέον είναι οι ε, εγκαυματίες με βαριά εγκαύματα μετά την πυρκαγιά αυτή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί σε αυτά τα ιδρύματα και κανείς δεν αναλαμβάνει παρόλες προειδοποίησεις. Η επόμενη στρατηγική αναπηρία δεν μπορεί να είναι ένα κενό γράμμα ή ένα έγγραφο για να το κοιτάξει το κράτο μέλο, να το βάλει σε ένα σιρτάρι και μετά να συνεχίσει να αγνοεί την κατάσταση. Χρειάζεται μια στρατηγική προσέγγιση. Ε, δεν υπάρχει σωστή καθοδήγηση στα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει ανταλλαγή καλών πρακτικών. Ένα άλλο σημαντικό στο έργο μας είναι να επικρίνουμε τα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν σωστά την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Αναπηρία, παρόλο που την έχουν κυρώσει. Υπάρχει αυτή η Σύμβαση του ΟΗΕ, ωραία, δεν εφαρμόζεται όμως ε, σε στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό να το λέμε. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε την κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να βοηθούμε και να γίνει μια ένωση, λέμε, που να μην αφήνει κανένα στην άκρη. Και, δεν συμπεριλαμβάνουμε αυτή τη σύμβαση του ΕΕ στι πολιτικέ μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει συστάσεις μετά στα κράτη-μέλη, τα οποία κράτη-μέλη συνεχίζουν να τις αγνοούν. Ε, και τελικά δεν υπάρχει φως για τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία μας, που είναι τα άτομα με αναπηρίες. χαμένη ευκαιρία. Είναι η ε, ε, πράξη για την ε, προσβασιμότητα. Στις μεταφορές και στα οχήματα η κατάσταση είναι χάλια. Καμιά φορά πηγαίνουν στα ιδρύματα τα ευρωπαϊκά κονδύλια και έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα λόγω της κακής συνεργασίας και συντονισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζει τη σύμβαση, τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τις συστάσεις, αδιαφορούν οι πάντες. Uh, member states Όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν ε, τα κονδύλια. what they use it. Αλλά δεν ξέρουμε πώς και γιατί. Πώς είναι δυνατόν μετά από 15 χρόνια συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε τέτοια ιδρύματα τεράστια γεμάτα άτομα με αναπηρία, με, με εκτρές συνθήκες. Μα πώς είναι δυνατόν αυτό. Measuring the Θα πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε τα αποτελέσματα. Ε, ε, όχι γενικά και αόριστα που πηγαίνουν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα. Στο ψήφισμα έχω τονίσει ότι η νέα στρατηγική για την αναπηρία θα πρέπει να έχει στόχους συγκεκριμένους, φιλόδοξους και ένα χρονοδιάγραμμα ή περισσότερα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή και όχι γενικολογίε και τα κράτη-μέλη που δεν ακολουθούν τις συστάσεις, τι πολύ συγκεκριμένες συστάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να τιμωρούνται κάποια στιγμή, να σταματούμε να τους χορηγούμε κονδύλια. Πρέπει να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Τι γίνεται όταν αδιαφορεί μια κυβέρνηση. Θα πρέπει να έχει συνέπειες. με τη σωστή χρηματοδότηση και το σωστό έλεγχο. Απολύτως απαραίτητα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. Ας είμαστε φιλόδοξοι και ας καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εγκαταλείπει ε, τους αναπήρους μας. Γιατί πραγματικά αυτοί έχουν την ανάγκη μας, δεν μπορούμε να τους παραμελούμε. Θα ακολουθήσει σύντομη ανταλλαγή απόψεων, αν μου επιτρέπετε. E από τους συντάκτες του ψηφίσματος, τους συνεισηγητές, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Κιμπουρόπουλος, παρακαλώ, και ζητώ συγγνώμη. Thank you, Mrs. Chair, and uh, thank you Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την ομάδα μου που μου ανέθεσε αυτή την ευθύνη. Θα μιλήσω ελληνικά. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που συζητάμε αυτό το ψήφισμα. Ε, κυρία Πρόεδρε, γραμματής, πραγματικά έχετε κάνει μια πολύτιμη δουλειά ε, με το προσχέδιο αυτού του ψηφίσματος που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό ε, αυτά που ακούστηκαν στην Ολομέλεια τον ε, προηγούμενο Δεκέμβριο στη διάρκεια της προφορικής ερώτησης που ε, ανέβασε και ε, ξεκίνησε το ΕΛΚ. Μιλάμε για ένα μη συγκρουσιακό θέμα, οπότε ας επιδιώξουμε να συνεργαστούμε υπερκομματικά σε αυτές τις τοπολογίες Αυτό θα ήταν πραγματικά μία πρόκληση. Μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Ε, στο ψήφισμα βλέπω τρεις προκλήσεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να μην, να δημιουργήσουμε ένα μακροσκελές ε, ευχολόγιο που στο τέλος θα χάσει την ουσία του. Όπως ε, πολύ καλά είπε και ο συνάδελφος και ο Σάνταμ Κόζα, πρέπει να μικρύνουμε και να το κάνουμε πολύ στοχευμένο ε, αυτό το, το κείμενο. Ακόμα και να διαγράψουμε κομμάτια είναι τροπολογία. Το δεύτερο στόχος είναι να είμαστε ξεκάθαροι. Για να μας ακούσει η Επιτροπή, στην, ε, το, ε, η Επιτροπή πρέπει να, να ε, να πρέπει να είμαστε σαφείς και πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη πενταετία. Ας δούμε τι δεν λειτουργεί. Ναι, έχουμε την Accessibility Act και έχει γίνει mainstreaming σε τόσο κείμενα, όμως το θέμα είναι, τηρείται, ε, έχει πρακτικότητα στην καθημερινή ζωή μας. Είναι θέματα που πρέπει ε, να δούμε και έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε σε αυτό το κείμενο. Προσωπικά προτείνω να δώσουμε έμφαση σε κάποια ζητήματα. Απασχολησιμότητα, κίνητα για εργασία, τόσο στο, στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, εκπαίδευση και πώς η τεχνολογία μπορεί να μπει στη ζωή μας, στη ζωή των ανάπηρων πολιτών και πραγματικά να βοηθήσει από όλες τις μεριές. Ζούμε, θεωρώ, σε μια εποχή που, ναι, η αναπηρία έχει δημιουργηθεί από την κοινωνία, αλλά η τεχνολογία μπορεί να στηρίξει και να εξομαλύνει αυτή την κατάσταση θεωρώ ότι πρέπει να τονίσουμε, γιατί είμαι και εγώ ένας άνθρωπος που δεν πιστεύω σε αυτή την πολιτική, ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα και μια πολιτική που χρειαζόμαστε, που, που θεσπίζουμε λιγότερα επιδόματα. Πρέπει οι άνθρωποι, οι ανάπηροι πολίτες να βγουν έξω στην κοινωνία και να, να, να, να, να παλέψουν και να έχουν τα εργαλεία για να παλέψουν όπως παλεύει ο κάθε πολίτης. Ε, πρέπει επίσης να μείνουμε σε κάποιες ειδικέ κατηγορίες όπως είναι οι γυναίκες, οι γυναίκες με αναπηρία. Θέμα που σηκώνει η κυρία Ρόζα Εσταράς. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε μέσα σε, αυτές τις, μέσα σε αυτή την τροπολογία ε, συνθήκες και εξειδικευμένες. Σας ευχαριστώ πολύ και πιστεύω και ε, είμαι εδώ για να κάνουμε έναν γόνιμο διάλογο. Thank you very much. The next one would be, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ένισελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην εισήγησή σα σωστά υπογραμμίσατε τη σημασία του θέματος και νομίζω πως μιλήσατε και για τις κύριες ε, προκλήσεις. Ε, σας ευχαριστώ για αυτό. Θέλω να ξεκινήσω, θυμίζω ότι έχουμε 80 εκατομμύρια ε, κόσμο στην Ευρώπη που ζει με αναπηρίες και τα 46 εξ αυτών είναι γυναίκες. Το 2016 υιοθετήθηκε ε, ε, μάλλον, ε, συγγνώμη, νωρίτερα υιοθετήθηκε η στρατηγική σχετικά με τους ανθρώπους με αναπηρίες για το 2010 μέχρι το 2020 και προήλθαν όλα τα στοιχεία αυτά από την σχετική έκθεση του ΟΗΕ το 2017 θα ήθελα λοιπόν να αναζητήσουμε μια γενική αναθεώρηση όλων των νομοθετημάτων της Ένωσης με βάση ε, τις συστάσεις CRPD του ΟΗΕ. Χρειάζεται δε επιβολή και εφαρμογή. Χθε είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Μερσή να συζητήσουμε το θέμα. Επίσης είναι σωστό ε, να υπογραμμίσουμε την ε, Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αναπτύξατε και εσείς αυτό, με κονδύλια, να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι οι ευρωπαϊκά κονδύλια δεν θα συμβάλλουν στην κατασκευή ή στην ε, ανακαίνιση ιδρυμάτων. Επίσης είναι σημαντικό να εγκρίνουμε το ε, ε, προαιρετικό πρωτόκολλο της σύμβασης ε, RPD και θέλουμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις, να δώσουμε περισσότερα αποτελέσματα, να εναρμονίσουμε τον ορισμό της αναπηρίας, της πρόσβασης και χρειάζεται φυσικά κοινωνική ασφάλιση, προστασία του εισοδήματος, κονδύλια για κοινωνική ένταξη, κονδύλια να μην δαπανώνται σε άχρηστες υποδομές ή υποδομές που θα ε, ε, αποτελούσαν διακρίσεις ενάντια στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Χρειάζεται επίσης να δουλέψουμε για μια ευρωπαϊκή κάρτα αναπήρου ε, και ειδικού χώρου στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίε σε ολόκληρη την Ένωση. Συνεργασία μου ως συνεισηγητής επίσης θα προσέξω πάρα πολύ τις συστάσεις που λαμβάνουμε από την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά ανοιχτοί προς την κοινωνία των πολιτών. Είχα ήδη ε, καλή συνεργασία με τους συναδέλφους στην ομάδα και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία με τους συνεισηγητές από τις άλλες πολιτικές ομάδες επίσης και θα μπορέσουμε έτσι να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Επιτροπή όταν ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τώρα την κυρία Μάξοβα εξ ονόματος των Πρασίνων, αλλά δεν είναι... Ρινιού. Του Ρινιού, συγγνώμη, αλλά δεν είναι ακόμα εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω γαλλικά η κυρία Μπρουνέ. Όντως για το Renew πρόκειται για ένα μείζονο σημασίας θέμα, το σχέδιο δηλαδή που θέλουμε να προτείνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινοβούλιο και Κομισιόν για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, αναπηρίες. Ειδικά στο χώρο της εργασίας θα πρέπει αυτό το μέσο να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσαρμοστούν κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο οι θέσεις εργασίας για να διευκολύνουμε την ένταξη των ανθρώπων αυτών. Επίσης, ιδιαίτερη επαγρύπνηση και το είπαμε για τις γυναίκες με αναπηρία μέσω της Επιτροπής των Γυναικών, όπου εγώ είμαι αναπληρωματικό μέλος, εργάζομαι για το θέμα των αποκλήσεων των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και θα ήθελα να το κοιτάξουμε ακόμα πιο προσεκτικά για τις γυναίκες με αναπηρία, όπου η απόκληση είναι ακόμα πιο μεγάλη, δηλαδή είναι διπλή διάκριση, διπλή επιβάρυνση για ε, είναι ε, διακρίσεις οι οποίες σωρεύονται ενάντια στις γυναίκες. Πρέπει αυτά τα κονδύλια λοιπόν να τα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε θέσεις απασχόλησης που συχνά είναι λιγοστές. Έχουμε το θέμα μας απασχολεί στη Γαλλία ακόμα και αν υπάρχουν υποχρεωτικά ε, ποσοστώσεις 6% προσωπικού σε ανθρώπους με αναπηρία που, που είναι υποχρεωτικό για τις εταιρείες ε, αλλά τα κονδύλια δεν είναι προσαρμοσμένα για κάθε φορά που πρέπει να προσαρμοστεί μια θέση απασχόληση σε άνθρωπο με αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Λάγκεν Ζήπεν. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Δεκέμβριο ε, ζήτησα από πλευρά των Πρασίνων να κάνουμε ένα ψήφισμα για τη στρατηγική αυτή μετά το 2020. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη συνέχιση της σημερινής στρατηγικής για την αναπηρία. Είναι θλιβερή πραγματικότητα ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες θερούνται των βασικών θεμελιωδών τους δικαιωμάτων παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα κράτη-μέλη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία. Η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι χιλιάδες ατόμων με αναπηρίες αναγκάζονται ακόμα να ζουν ε, ε, έγκλειστοι σε ε, ιδρύματα χωρίς ευκαιρία να συμμετέχουν στην κοινωνία και με απάνθρωπες συνθήκες. Να σταματήσουμε εδώ, να σταθούμε και να τιμήσουμε αυτούς τους οχτώ ανθρώπους με πνευματική αναπηρία που έχασαν τη ζωή τους σε μια ε, πυρκαγιά ε, ε, στην Τσεχία σε ένα υποτιθέμενο ίδρυμα εντός εισαγωγικών. Θα πρέπει να απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους οι άνθρωποι με αναπηρίες και να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή. Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τη στρατηγική μας μετά το 2020, γιατί στρατηγική χρειαζόμαστε, αλλά να καλύπτει όλες τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, που να έχει φιλόδοξους στόχους ε, και χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή που να συμπεριλαμβάνονται απολύτως ε, στο πλαίσιο διακυβέρνησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική ακριβώς με ειδικού στόχους που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα ε, των ατόμων με αναπηρία που μπορεί να είναι και θύματα διακρίσεων σε όλες τις πολιτικές. Αυτή η μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να καταρτιστεί με συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων τους των αντιπροσωπευτικών και να συμμετέχουν συνέχεια στις διαβουλεύσεις ε, στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την εποπτεία της Επιτρόπου Ντάλη. Θα πρέπει συστηματικά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να μπαίνουν σε όλες τις πολιτικές, ε, στην νομοθεσία, στα προγράμματα, ε, ακόμα και στην πολιτική ισότητα του φίλου, Με ιδιαίτερη προσοχή επίσης και στην καταπολέμηση της βίας και στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Περιμένουμε πολλά από αυτή την Task Force για την ισότητα, αλλά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να καταρτιστεί μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη στρατηγική για την περίοδο μετά το 2020. Ευχαριστώ για να κλείσει ο κύκλος των συντακτών ε, θα πάρει το λόγο η κυρία Ραφάλσκα και μετά τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα από την αρχή να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη και σας ευχαριστώ για το ψήφισμα αυτό. Ακούσαμε και από τους προλαλήσαντες ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα για όλους μας. Αυτή η νέα στρατηγική χρειάζεται φιλοδοξία, αλλά και ε, αντικειμενικότητα και νυφανιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τις πιο ανεπτυγμένες και από τις πιο πλούσιες ε, περιοχές στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά παραμένουν ακόμα πολλοί πολίτες της Ένωσης, πάνω από 80 εκατομμύρια, ε, που αισθάνονται ή είναι όντως αποκλεισμένοι από την κοινωνία. Χάνουμε πολύτιμες δεξιότητες, πολύτιμες ικανότητες, γιατί τα άτομα με αναπηρία δεν βρίσκουν το δρόμο τους στην αγορά εργασίας δυσκολεύονται πολύ. Η στρατηγική μετά το 2020 είναι απολύτως απαραίτητη ακριβώς ε, για να καταλάβουμε ότι ε, τα άτομα με αναπηρίες είναι αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας μας. Πρέπει οπωσδήποτε να ε, βρούμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση. Γιατί όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε για να εφαρμοστούν χρειάζονται χρήματα. Ε, χρειάζεται χρόνος ε, σωστά χρονοδιαγράμματα και καλή παρακολούθηση και έλεγχος για το πώς υλοποιούνται όλα αυτά. Οι διαβουλεύσεις είναι πολύ σημαντικές στο κοινωνικό διάλογο ε, για την εκπόνηση της νέας στρατηγικής. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται επίσης σωστά με τρόπο πολύ κατανοητό και ε, για τα άτομα με αναπηρίες και καλά οργανωμένο. Επίσης θα πρέπει να συμμετέχουν στην εκπόνηση και οι ίδιοι με τις οργανώσεις τους. Περιμένουμε από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να αντιδράσουν. Η συγκήτριά μας, η πρόεδρος, τόνισε ότι πρέπει να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα. Ε, είναι απολύτω απαραίτητη αυτή η στρατηγική. Πρέπει να συνεχιστεί ε, με τρόπο αποτελεσματικό, φιλόδοξο. Είναι 8 πολύ συγκεκριμένοι τομεί δραστηριοτήτων και δεν θα πρέπει να τους ξεχνάμε. Παιδεία, εκπαίδευση, κατάρτιση, υγεία, προστασία της κλπ. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, η Πρόεδρος. Μάλιστα, θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Κώσε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας συγχαρώ για την πρόταση αυτή. Ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολύ καλή ε, δουλειά και πολλή δουλειά. Έχω διατελέσει κι εγώ εισηγητής ε, στην πρώτη μου θητεία για το θέμα αυτό. και συμμετείχα και στην εκπόνηση της προηγούμενης στρατηγικής μέχρι το 2020. Υπάρχει ένα ζήτημα με την κινητικότητα των προσώπων με αναπηρίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό οι μετακινήσεις. Ε, υποτίθεται γενικά ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας, ε, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να συνεχιστεί η στρατηγική μετά το 2020. Παραμένει πολλή δουλειά, ό,τι και να έχουμε πετύχει. Είναι πολλά τα εμπόδια, πολλές οι δυσκολίες και έχουμε και πολύ καλές προτάσεις όμως για τη λύση και με την ψηφιοποίηση. Και επίσης αυτό βοηθάει για την ουσιαστική ένταξη ε, στην κοινωνία και στην εργασία των ατόμων με αναπηρίες. Πρέπει οπωσδήποτε το διάστημα μετά το 2020 να υπάρχει μια ε, σωστή στρατηγική, στοχευμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική. Με γνώμονα ε, τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με χρειάζεται οπωσδήποτε να βασιστούμε στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και να εφαρμόσουμε όλα τα σημεία. Η χρηματοδότηση επίση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όπως ακούσαμε, γιατί αυτή τη στιγμή όλα αυτά χωλένουν. Ε, άκουσα πρόσφατα ότι το τελευταίο διάστημα πολλά από τα έργα τελικά ε, δεν ολοκληρώθηκαν, δεν υποστήριξαν τους ε, δικαιούχους δεν συμμετείχαν οι δικαιούχοι και τελικοί αποδέκτες στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση και τελικά υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ που πηγαίνουν στην έρευνα, που πηγαίνουν σε διάφορα έργα και προγράμματα ερήμην των ε, προσώπων με αναπηρία που αυτοί ξέρουν καλύτερα τι χρειάζονται. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και τους ε, φραγμούς παντού σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να σας επιστήσω την προσοχή σε κάτι ακόμα. Έχω ξαναπεί σε πολλές συζητήσεις ε, ότι θεωρώ πολύ μεγάλο πρόβλημα τις διακρίσεις κατά των ε, προσώπων με αναπηρίες. παραμένουν οι διακρίσεις και είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει νομίζω να το ξανασκεφτεί και να προσπαθήσει να προτείνει καλύτερες λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει και ακυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Δική μας ευθύνη τώρα είναι να δώσουμε συνέχεια και να σταματήσουν οι διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες. Uh, Τώρα, κυρία Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την Προεδρία Πράγματι η στρατηγική αυτή ε, χρήζει εμβάθυνσης και περαιτέρω εξέτασης. Έχουμε καταθέσει ορισμένες τροπολογίες που στόχο έχουν τη διεύρυνση θα έλεγα ε, της συγκεκριμένης πρότασης. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους θα πρέπει να εμείνουμε όπως η ισότητα, η συμμετοχή, ε, ο κοινωνικός αποκλισμός και η καταπολέμησή του και φυσικά η υγεία. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τους ανηλίκους, με τους νέους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν επιπλέον θέματα. Και να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ενηλίκους και θα πρέπει να ε, επιτρέψουμε στα παιδιά να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτά. Έχει επίσης μεγάλη σημασία να κάνουμε αναφορά στην ανάγκη που υπάρχει να γίνουν διακρίσεις ανάμεσα στις αναπηρίες και αν είναι σωματικές, αν είναι διανοητικές και ε, να υπάρξουν έτσι ειδικότερα μέτρα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες ε, κάθε ε, θα έλεγα κατηγορίας. Συνεπώς λοιπόν Υπάρχουν επίσης και τα θέματα των συνδυασμών αναπηριών, υπάρχουν τα θέματα των κοφαλάλων σαν παράδειγμα που ταυτόχρονα έχουν και προβλήματα όρασης και για αυτές τις κατηγορίες που φύγονται από δύο αναπηρίες θα πρέπει να υπάρξουν πιο συγκεκριμένα μέτρα. Ένα άλλο θέμα είναι η συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία στην οικονομία, στις οικονομικές δραστηριότητες αλλά και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε η κυρία Φράνσεν. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη πρόταση. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει συνεκτικότητα στο εσωτερικό του πυλώνα του Ευρωπαϊκού για τα κοινωνικά δικαιώματα. Κάποια σημεία. Καταρχάς θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει πραγματικά τα ευρωπαϊκά κράτη στον τομέα της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα θα πρέπει να υπάρξει επίσης στοχευμένη βοήθεια του Κοινωνικού Ταμείου στον τομέα της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας. Και όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν φυσικά και στις προβλέψεις της δημοσιονομικές για τα θέματα της αναπηρίας. Μαρίνο. Συμφωνώ πλήρως, λέει ο κύριος Μαγιορίνο, με την κατεύθυνση την οποία έχει πάρει η συζήτηση και θα ήθελα να θυμίσω ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, έχουμε ένα βασικό μέσο στη διάθεσή μας, είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε σαν μια σταθερή σιωπηλή, ίσως αλλά σταθερή και μόνιμη ε, πλατφόρμα αναφοράς σχετικά με την ανάπτυξη των πολιτικών τις οποίες θα αποφασίσουμε. Δεύτερον, κάθε συζήτηση για τα θέματα των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία θα πρέπει να είναι στα πλαίσια ενός διαλόγου με τους πολίτες με αναπηρία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε όλες τις δυνατότητες ανοιχτές έτσι ώστε να συμμετέχουν άμεσα οι άνθρωποι στους οποίους αφορά η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Ένα τρίτο θέμα. <coughs> Μιλάμε για ανθρώπους με αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για κάποιες συνθήκες οι οποίες μεταξύ τους είναι διαφορετικές. Έχει σημασία λοιπόν η λεγόμενη προσωποποίηση των προτάσεων αυτών έτσι ώστε οι δυνατότητες να καλύπτουν τις διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές προελεύσεις, διαφορετικές παθολογίες και τελικά διαφορετικές ανάγκες. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει κάποιες γενικές προτάσεις και προσπάθειες να κάνουμε όπως η αυτονομία ε, το θέμα των γυναικών, το θέμα της φτώχειας, φυσικά όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ απαιτητικοί σε σχέση με την βοήθεια που δίδεται στις περιπτώσεις ε, θα έλεγα υψηλών αναγκών. Να μην κάνουμε το λάθος, να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, είναι κάτι το οποίο θα καλυφθεί από την εξειδίκευση των πολιτικών αυτών από τα κράτη-μέλη. Τα τελευταία χρόνια είδαμε στην Ευρώπη να ακολουθούνται καταστάσεις και πολιτικές οι οποίες μεταξύ τους διαφοροποιούνται εντελώς. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει από τη μία να διευκρινίσουμε τους στόχους και από την άλλη όμως να καθορίσουμε κάποια επίπεδα απαιτήσεων κάτω από τα οποία ποτέ δεν θα πρέπει κανένα κράτος μέλος να κατεβαίνει στον τομέα των αναπηριών. Πρέπει να είμαστε απαιτητικοί λοιπόν και στον τομέα των επενδύσεων και θα πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί και σε σχέση με τις κυρώσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου εξέφρασε αρκετές προτάσεις οι οποίες ε, είναι πολύ σωστές και πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες οι οποίες όμως δεν έχουν καταστεί ακόμα τμήμα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει λοιπόν αυτό να το διευκρινίσουμε. Mr. and then Madame Ehm, najlepša hvala eh, za besedo. Eh, tudi sam eh, pozdravljam resolucijo. Και εγώ θεωρώ ότι η πρόταση αυτή είναι μια θετική πρόταση. Θα πρέπει καταρχάς να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. έχει μεγάλη σημασία ε, εδώ βέβαια το πώς βλέπουμε γενικότερα τα δικαιώματα των πολιτών. Πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν την χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οποία δυστυχώς ε, θυμίζω ότι ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε ακόμα επικυρώσει, για λόγους στους οποίους είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε τις απαιτήσεις αυτής της χάρτας να τις μεταφέρουμε στις δικές μας ε, νομικές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερα όταν τίθενται θέματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός. Γι' αυτό λοιπόν η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού για τους συμπολίτε μας με αναπηρίες είναι μια προτεραιότητα μαζί με την καταπολέμηση της φτώχειας κτλ αλλά θα πρέπει να γίνει εδώ μια διάκριση ανάμεσα στην κατάσταση η οποία συνεισφέρει και οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό και στις προσπάθειες τις οποίες πρέπει να κάνουμε εμείς για την αυτονομία των συμπολιτών μας με αναπηρίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει και αναχώρα, αλλά θα πρέπει να γίνει και με συνεργασίες ανάμεσα στις χώρες όπου εκεί είναι χρήσιμο. Ε, για την αυτονομία στην ζωή των συμπολιτών με αναπηρίες ε, θα πρέπει να διευκρινίσουμε λίγο και τις ανάγκες ε, τις οποίες έχουν τα οικογενειακά πλαίσια μέσα στα οποία βιώνουν οι άνθρωποι με αναπηρίες πέρα από την βοήθεια την οποία παίρνουν από τους οργανωμένους ε, ε, θα έλεγα μηχανισμούς, κρατικούς, κοινωνικούς κτλ πρέπει να καθοριστεί και η βοήθεια προς τους οικογένειες οι οποίες φροντίζουν τους συμπολίτε μας αυτούς. Μπίσοφ και εγώ. Θα ήθελα να πω ότι ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα κοινωνικό πυλώνα, πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η ισότητα των ευκαιριών για όλους. Και ρητά να λέμε ότι ε, ε, αυτό αφορά και τα άτομα με αναπηρίες. στο κείμενο διαπιστώνεται αυτό, το γράφει ήδη δηλαδή, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό από την ευρωπαϊκή σκοπιά όχι μόνο από την εκάστοτε εθνική σκοπιά στα κράτη-μέλη. Βλέπω όλο και περισσότερο και ακούω ανθρώπους που έρχονται και μας λένε τα βιώματά τους και τις εμπειρίες τους. Στη Γερμανία υπάρχει να ταυτότητα ε, που τους εξασφαλίζει πρόσβαση σε διάφορα πράγματα και μετά πηγαίνουν διακοπές σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και δεν τους αναγνωρίζεται τίποτα. Τώρα είμαστε στο έτος 2020 και δεν τα έχουμε ακόμα καταφέρει και αυτό είναι πραγματική ντροπή. Ε, θα πρέπει να πιέσουμε και να πούμε ότι θα υπάρξει μια κάρτα είτε πανευρωπαϊκή ταυτότητα ή τουλάχιστον αναγνωρίζεται η εθνική και στα άλλα κράτη-μέλη. Για να μην ε, αντιμετωπίζει ο κόσμος τέτοια τεράστια προβλήματα όταν ξαφνικά κάπου πηγαίνει διακοπές. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, επειδή στη Γερμανία είναι πολύ επίκαιρο. Έχουμε πάνω από 300.000 ανθρώπους που εργάζονται σε σχετικά εργαστήρια και υπάρχει μελέτη του Υπουργείου Εργασίας πριν από 2-3 χρόνια και ε, ο μισθός, η αμοιβή τους είναι κατά μέσο όρο, παρακαλώ, 180 ευρώ το μήνα. 180 ευρώ. Έχουν κανονικό 35 ώρο. Πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά. 1,3 ευρώ την ώρα βγαίνει. Είναι και αυτό απαράδεκτο και κάτι πρέπει να τα αλλάξουμε και όχι ωραίες ομιλίες να βγάζουμε και κηρύγματα, να συμμετέχουμε στην κοινωνία και να αλλάζουμε τα πράγματα. Και όχι απλώ να αξιολογούμε και να εκτιμούμε τη δουλειά τους, να την αμείβουμε και όλα σωστά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα θέλαμε τώρα να ακούσουμε κάτι και από πλευρά Κομισιόν. Madame Placencia Porero. Yes, hi, sorry. Thank you. Um, σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για το σχέδιο ψηφίσματος που διαβάσαμε με μεγάλη προσοχή και για τα σχόλια που κάνατε σήμερα. Όπως είδατε από την ανάληψη καθηκόντων του Επιτρόπου, της Επιτρόπου Ντάλη, είναι μια προτεραιότητα ε, οι άνθρωποι με αναπηρία για την καινούργια επιτροπή. Θα δοθεί μεγάλη προσοχή σε αυτό το θέμα και για να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας θα θέλαμε να παραπέμψουμε στο πρόσφατο ανακοινωθέν που υιοθετήθηκε σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων όπου επιβεβαιώνεται ότι μια ενισχυμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για του ανθρώπου με αναπηρία θα ε, προταθεί ότι το 2021 αναγνωρίζει τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία ακόμα σήμερα στην Ευρώπη και προετοιμάζοντας αυτή τη στρατηγική, οι συμβολές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι φυσικά πολύ ευπρόσδεκτες. Στην προετοιμασία λοιπόν αυτή τη ε, νέα στρατηγική ε, βλέπουμε μια καλή ευκαιρία για να προωθήσουμε την κύρωση τη σύμβαση και αυτό μα βαραίνει με ευθύνε ώστε να εξασφαλίσουμε πω οι άνθρωποι με αναπηρία θα έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που αναγνωρίζει η σύμβαση αυτή. Είμαστε καλύτερα τώρα εξοπλισμένοι από ό,τι πριν 10 ε, χρόνια όταν παρουσιάσαμε την προηγούμενη στρατηγική γιατί επιτύχαμε αρκετά αποτελέσματα που μας βοηθούν στην πρόοδο. Έχουμε περισσότερα δεδομένα, έχουμε ε, νομοθεσία, έχουμε δαπανίσει τα κονδύλια, πράγμα που μας κάνει να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά και να ε, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τις φιλοδοξίες όλες αυτές, ε, να τις μετατρέψουμε σε πράξη. Επίσης θα έχουμε πληροφορίες από την αξιολόγηση της ε, ισχύουσας στρατηγικής που έχει ήδη προχωρήσει αρκετά και έχουμε εξετάσει πολύ προσεκτικά τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για αξιολόγηση που ήδη περιλαμβάνει κάποια στοιχεία ε, για τις κύριες ανησυχίες ε, και προβληματισμούς που έχουν ε, οι άνθρωποι με ειδικέ ανάγκες. Εμείς δουλεύουμε με τους ανθρώπους με αναπηρία και τους εκπροσώπους τους για να προετοιμάσουμε τη στρατηγική μετά το 2020. Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά και την τελική εκδοχή της έκθεσης με όλες τις τροπολογίες που θα υποβάλλετε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο 23 την ε, παρουσίαση της κατάστασης ΡΟΑΔΟ όσον αφορά το, ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπλίνκεβιτσούτε που είναι η συγγήτριά μας. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εχθές στην ε, Επιτροπή μας μιλήσαμε για την έναρξη διαπραγματεύσεων διοργανικών και τα ψηφίσαμε κιόλα. Περιμένω λίγο. E, e, Συνεχίζω. Χτες ε, έγινε μια ψηφοφορία στην Επιτροπή, έλεγα, για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ήδη για τον τριμερή διάλογο. Η πρώτη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 4 Φεβρουαρίου. Είμαι η Και θα ήθελα να σας θυμίσω τη θέση μας από την πρώτη ανάγνωση, από τις πρώτες διαβουλεύσεις και ποια είναι τα σημαντικά για μας. Αυτό το ταμείο είναι ταμείο αλληλεγγύης. Βοηθάει τους απολυμένους να ε, μετεκπαιδευτούν, να καταρτιστούν, να βρουν άλλη δουλειά κτλ. Έτσι ώστε όσοι έχουν χάσει την εργασία τους να μπορέσουν να επανέλθουν γρήγορα στην αγορά εργασίας και να βρουν δουλειά αυτό είναι πραγματικά ε, ένα κοινωνικό ταμείο για τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους. Από το 2006 έχει αρχίσει η εφαρμογή του και κανονικά στόχο έχει να βοηθήσει τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους και απολύονται λόγω παγκοσμιοποίησης μετεγκατάστασης ε, των επιχειρήσεων που δούλευαν κτλ. Μετά ήρθε να προσθεθεί και η ε, χρηματοοικονομική κρίση. Να βοηθήσουμε τους νέους ε, που δεν είναι σε εκπαίδευση, σε κατάρτιση, σε μαθητεία. Ιδιαίτερα στις περιφέρειες ΝΑΤΣ 2. Τώρα καλούμαστε να αποφασίσουμε πώς θα ενταχθεί αυτό το ταμείο στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Τι στόχο θα έχει και πώς θα ε, λειτουργήσει στο μέλλον. Έχει καταθέσει μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου Μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων ανά εταιρεία από 500 σε 250 για να είναι επιλέξιμη. Ε, είναι πολύ πιο απλή η διαδικασία ε, και οι προθεσμίες. Όλα αυτά ωραία. Στις 16 Ιανουαρίου πέρσι μάλλον φέτος στις 16 Ιανουαρίου εμείς ε, διατρονώσαμε τη δική μας θέση που είναι ακόμα πιο φιλόδοξη από εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. για να είναι πιο αποτελεσματικό στη στήριξη ε, των απολυμμένων. Τα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή και να προσθέσουμε ε, να ληφθούν υπόψη και οι τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση, Brexit κλπ. Γιατί αυτό είναι που ε, διωγγώνει την ανεργία. E ε, γι' αυτό λοιπόν ο στόχος μας είναι τα μέτρα και τα μέσα να αποφασιστούν ε, πολύ ε, συγκεκριμένα με βάση το σκοπό της, της ε, υπόθεσης αυτής του Ταμείου και όχι τα αίτια, δηλαδή όχι γενικά την παγκοσμιοποίηση, αλλά πού θέλουμε να φτάσουμε, σε ποια αναδιάρθρωση και θέλουμε να μειώσουμε και τον αριθμό των εργαζομένων στους 200 από τους 250 που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχικά ήταν 500, θυμίζω. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να πάρουμε ενεργά μέτρα και να περιλαμβάνουν και την πρόνοια για τα παιδιά. Θα πρέπει οπωσδήποτε τα παιδιά των εργαζομένων αυτών να εξασφαλίζονται, να ε, υπάρχει μέρημνα για τη φροντίδα τους, για να μπορούν οι γονείς να ασχοληθούν με την εξέβρεση εργασίας και την αναζήτηση, κατάρτιση, εκπαίδευση, να ξέρουν ότι τα παιδιά τους είναι κάπου για να μπορούν οι ίδιοι να ε, ψάχνουν για δουλειά. Και ε, να διατηρηθεί και χρηματοδότηση για τους νέους Επίσης θέλουμε μία άπαξ καταβολή 20 με 25 χιλιάδων ε, για κάποιους που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Ε, να ανοίξουν τα βιβλία τους, ένα εφάπαξ, ας πούμε, μια μαγιά 20 με 25 χιλιάδες. Επίσης, κάτι άλλο που μας προβλημάτισε είναι και ο ίδιος ο τίτλος ε, του Ταμείου. Για να ανταποκρίνεται καλύτερα στο σκοπό και στο στόχο του Ταμείου. Ελπίζω να τα βρούμε τελικά με το Συμβούλιο και να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, εμείς δεν θα ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή με τα πολιτικά ζητήματα μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο για το τελικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πραγματικά ε, θα είμαι πολύ αυστηρή σε αυτό. Θα συμμετέχουμε φυσικά και εμείς στις ε, διαπραγματεύσεις, αλλά αν δεν έχουμε τελικά αριθμητικά στοιχεία και ποσά ακόμα από το Συμβούλιο για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στους τριμερείς διαλόγους συζητάμε μόνο τα τεχνικά ζητήματα και όχι τα οικονομικά. Ε, θα συζητήσω λοιπόν με τους κοιόδης ηγητές. Στις 4 Φεβρουαρίου είναι η συνεδρίασή μας και θα δούμε ε, πώς θα ε, διαμορφώσουμε την τακτική μας για τις διαπραγματεύσεις και το χρονοδιάγραμμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ε, μπορώ να καλωσορίσω ε, ε, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπλίνκεβιτσούτη και δίνω το λόγο στην κυρία Σουκόβα της Επιτροπής, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους, αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητή Συγγήτρια. Αγαπητοί ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ πολύ που προχωρήσατε χτες με την υιοθέτηση τη εντολή, πράγμα που μα δίνει να, τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε το τριμερή στι 4 Φεβρουαρίου, όπω ανέφερε και η κυρία Μπλινκεβιτσούτη. Είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε για όλα τα στοιχεία που είναι δυνατόν να συμφωνηθούν ε, σε αυτή την τελευταία χρονιά πριν ξεκινήσει η επόμενη προγραμματική περίοδος. Ε, ξέρουμε τι διαδικασίε του κανόνε όχι τα χρήματα γιατί Ακόμα ε, συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα στους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων. Τι είναι λοιπόν το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και πώς δουλεύει. Από την αρχή, από τη δημιουργία του το 2006 και το, από το 2007 που άρχισε πια να λειτουργεί, ε, έχει παίξει το πολύ σημαντικό ρόλο πέρα από τον προπολογισμό πλαίσιο για να στηρίξει ε, εργαζόμενους που έχασαν τις θέσεις τους, ε, κυρίως λόγω για ε, των αιτίων, που ανέφερε η κυρία Μπλινκεβιτσούτε, άλλαξε όμως και το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου. Πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους όταν αυτή η απώλεια μπορούσε να αιτιολογηθεί από την παγκοσμιοποίηση. Μετά όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το πεδίο εφαρμογής και οι παρεμβάσεις βασίστηκαν και στις επιπτώσεις της κρίσης στους ε, ε, ανθρώπους. Και τώρα έχουμε ε, ξανασκεφτεί το πεδίο εφαρμογή και το έχουμε επεκτείνει και στους νέους για την παιδεία τους όταν δηλαδή σκεφτήκαμε το πεδίο εφαρμογή ε, του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση, η Ευρώπη είχε να αντιμετωπίσει πρόβλημα με πολλού νέου που δεν ε, παρακολουθούσαν ε, ούτε κατάρτιση, ούτε ανώτατε σπουδέ, ούτε επαγγελματικέ σπουδέ και γι' αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε μέσα και από το Κοινωνικό Ταμείο να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη και περιφέρειες όπου οι απώλειες θέσεων απασχόλησης ήταν πολύ πολλές να μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε και τους νέους που δεν ε, παρακολουθούσαν κάποια εκπαίδευση. Όταν υπήρχαν μεγάλες ε, ανακατατάξεις σε κάποια περιφέρεια, οι ε, ε, ε, νέοι δυσκολεύονταν ακόμη περισσότερο να βρουν δουλειές. Από ό,τι φαίνεται τώρα τα πράγματα πάνε καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι παλαιότερα και γι' αυτό για την επόμενη προγραμματική περίοδο δεν έχουμε προτείνει την κάλυψη των νέων γιατί έχουμε συγκεκριμένη θεματική εστίαση από, υπό το Κοινωνικό Ταμείο για τη στήριξη των νέων και, αλλά και επειδή δεν θέλουμε να περιμένουμε να απολυθούν μαζικά σε κάποια περιφόρια και μετά μόνο να ασχοληθούμε με τους νέους στην περιφέρεια. Θέλουμε να ασχοληθούμε με τους νέους από την επόμενη προγραμματική περίοδο μέσω του Κοινωνικού Ταμείου. Έχουμε το 2019 ήδη εισάγει ε, κάποια μέτρα προφύλαξης, αν τα πω έτσι, ότι δηλαδή αν έχουμε Brexit άνευ συμφωνία, θα υπάρχει δυνατότητα να κινητοποιηθεί το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση και να στηρίξει περιφέρειες όπου ο αντίκτυπος θα είναι σοβαρός στην απασχόληση. Ανέφεραν εν συντομία και η κυρία Μπλινκιβιτσούτα το ανέφερε την αλλαγή στις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του Ταμείου. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 500 απώλειες θέσεις απασχόληση σε μία, σε μία εταιρεία ή σε συνεργαζόμενες εταιρείε σε μία περίοδο τετράμινη ή αυτές οι 500 απολύσεις θα μπορούσαν να γίνουν σε διάφορες εταιρείες, σε συγκεκριμένες μικρομεσαίες στον ίδιο τομέα και στην ίδια περιφέρεια ή σε δύο γειτονικές ε, περιφέρειες αλλά ε, σε μια χρονική περίοδο εννιάμινη. Και στην τωρινή προγραμματική περίοδο έχουμε αυτή την εξαίρεση για μικρές αγορές εργασίας και για ε, εξαιρετικές περιστάσεις όπου οι απολύσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, ακόμα και αν είναι κάτω από το όριο των 500 ανθρώπων. Οι δραστηριότητε και η κυρία Μπλίνκεβιτσούτα ανέφερε κάποιε απαιτήσει, κάποιου όρου για περισσότερη ευκρίνεια και ε, ε, όσον αφορά ότι το ταμείο αυτό κυρίως στηρίζει ανθρώπους, όχι εταιρείε και παρέχει ε, πρακτικά μέσα για την αγορά εργασίας όπως επανεκπαίδευση, ε, η βελτίωση των ε, προσόντων, βοήθεια προς τις νεοφυείς εταιρείες, κατάρτιση Ε, μέχρι 50.000 ε, μπορεί να δοθούν για ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν μια εταιρεία. Όπως είπα, είναι παθητικά μάλλον, συγγνώμη, παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας δεν προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν. Ε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε ανθρώπους που αναζητούν εργασία, που ξεκινούν κατάρτιση, που Δίνουμε δηλαδή ε, χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τέτοιου είδους μαθήματα ε, Πρόκειται για επιδόματα τα οποία λειτουργούν ως κίνητρα για να μπορέσουν να βοηθήσουν ανθρώπους να συμμετέχουν στις ε, στις δραστηριότητες αυτές. Ωστόσο, έχουμε ένα ανώτατο όριο μέχρι 35% της εφαρμογής του Ταμείου μπορεί η στήριξη να φτάσει μέχρι το 60% του συνολικού κόστους ανά περίπτωση εξαρτάται από το κράτος, την εθνική νομοθεσία, το υπόλοιπο χρηματοδοτείται από το κράτος, από την περιφέρεια, από τις τοπικές αρχές και από ιδιωτικά κονδύλια. Μπορεί δηλαδή να είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε εθνική ιδιαιτερότητα, κανόνες κτλ. Θα πρέπει μια, ε, ε, ε, κάθε περίπτωση, κάθε αίτηση να τίθεται σε εφαρμογή εντός 24 μηνών από την αίτηση. Δηλαδή δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε ακόμη περισσότερο την έναρξη αυτής της στήριξης που δίνεται στους ανθρώπους στη χώρα ή στην περιφέρεια, για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή ε, περνάνε 300 μέρες μέχρι να εγκριθεί το καθέτημα. Που δεν μετράνε όμως για την εφαρμογή. Αυτοί που στηρίζονται είναι οι εργαζόμενοι που έχασαν τη θέση τους στη διάρκεια της περίοδου αναφοράς και δεν διαφοροποιούμε ανάμεσα στα είδη συμβάσεων ή απασχόλησης που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να ήταν μόνιμοι υπάλληλοι, μπορεί να ήταν ορισμένου χρόνου, προσωρινή Ή μπορεί να συνδέονταν με τη λειτουργία μιας εταιρείας, δηλαδή να δούλευαν με κάποια συνδεδεμένη ε, μια συνδεδεμένη εταιρεία. Με συγχωρείτε, μήπως μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει η Πρόεδρος. Μάλιστα, θα προσπαθήσω. People Όπως είπα, πρόκειται και για εταιρείε συγγενικές, ε, ε, δηλαδή συνεργαζόμενες. Όλοι όσοι επηρεάζονται από την κατάσταση μιας μεγάλης εταιρείας, δηλαδή μπορεί να είναι ε, δικαιούχοι. Από τότε που ξεκίνησε την ε, εργασία του το EGF το 2007 είχαμε 160 ε, περιπτώσεις από 21 κατημέλη και έχουμε στηρίξει 150.000 εργαζόμενους και πάνω από 4.000 νέους που δεν, ήταν, δεν εργάζονταν ή δεν παρακολουθούσαν κάποια εκπαιδευτικά μαθήματα η επιμόρφωση. Τα σπουδαιότερα αποτελέσματα ήταν το 2009 με 2011, όπου είχαμε την πολύ δύσκολη οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο, όπως ξέρετε, στην οικονομία και ορισμένες εταιρείες. Έχουμε μία μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση το 2008. Ήταν αυτό μια από τις κύριες βάσεις για να επανεξετάσουμε την πρόταση και βασιστήκαμε σε αυτή την ε, αξιολόγηση πριν κάνουμε την ε, νέα μας πρόταση. Η μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση κατέληξε τα πορίσματα ότι έχει αποτελέσματα, επέκτηνε τις υπηρεσίες τους απολυμμένους εργαζομένους. Επίσης, οι παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού αυτού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης ήταν εμφανείς, γνώριζαν οι άνθρωποι ποιος και, τι, ε, τους, και πώς τους χρηματοδότησε. Επίσης έδειξε ότι το ισχύον ε, όριο δεν αρκεί γιατί η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει ευρύτερα τις οικονομικές δραστηριότητες μιας εταιρείας και πολλών εταιριών μάλιστα που είναι αλληλένδετες. Δεν μπορείς δηλαδή να διακρίνεις ξεκάθαρα ποιο είναι ο αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιοποίησης ή αν αντιμετωπίζει γενικά οικονομικές δυσκολίες η συγκεκριμένη εταιρεία και γι' αυτό αποφασίσαμε ότι πρέπει να διευρύνουμε τους ε, λόγους για τους οποίους μπορεί να γίνει μια τέτοια παρέμβαση και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην πρότασή μας. Έχουμε βιωσιμότητα, βιωσιμότητα ε, που ορίζεται στο EGF γιατί λέει ότι η ε, βοήθεια θέλει να ε, παροτρύνει στην αναζωογόνηση και προσαρμογή των ε, τοπικών δημόσιων υπηρεσιών εξέβρεσης εργασίας για να βοηθήσουν τον κόσμο που έχει χάσει τη δουλειά του. Τώρα η διάρκεια της διαδικασίας έχει επικριθεί ότι δεν είναι αποτελεσματική γιατί όπως είπα 300 μέρες μας παίρνει να εγκρίνουμε οπότε προτείναμε μια αναπλοποίηση της διαδικασίας για αυτό το σκοπό. Η πρόταση σύντομα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης είναι ένα ειδικό ε, μέσο εκτός των ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού θα εξυγχρονιστεί ακόμη περισσότερο. Έχουμε 170 εκατομμύρια. Εμείς προτείνουμε 245 τώρα ως ανώτατο όριο για το ταμείο αυτό έχουμε διατηρήσει τον τίτλο ω είχε Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, γιατί όπως ανέφερα είναι πολύ γνωστό ε, και ο κόσμος ξέρει ότι αυτό το μέσο το οποίο κινητοποιείται κεντρικά στοχεύει στις περιφέρειες, στις συγκεκριμένε ομάδες ανθρώπων που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω της αναδιάρθρωση μια εταιρεία ε, για πολλούς και διάφορους λόγους. και θα διατηρηθεί ως ένα ε, δημοσιονομικό μέσο που στηρίζει νέους ανθρώπους, δημιουργεί νέες ευκαιρίες, ε, ε, οποιοδήποτε είδος επιπλέον βοήθειας που μπορεί να ισχύσει γενικά εκτός του EGF θα ισχύσει και προτείνουμε να μειωθεί το κατόφλι στους 250 εργαζόμενους. Ξέρω πως η κυρία Μπλίνκεβιτζούτε ανέφερε το όριο 200 εργαζομένων που προτείνει το Κοινοβούλιο. Είδαμε πως οι μεγάλες εταιρείες, μάλλον όλο ένα και λιγότερες εταιρείες ξεκινάνε με τα ρυθμίσεις και μαζικές απολύσεις ενώ περισσότερο οι μισές εταιρείε αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του ανταγωνισμού και των απαιτήσεων για παγκοσμιοποίηση, ψηφιοποίηση. Γι' αυτό και προτείναμε τον, ε, το όριο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των 250 εργαζομένων. Ανέφερα και τους νέους που δεν ε, αποσχολούνται ούτε ε, παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα, γιατί αυτό αυτό, αυτό το μέσο βοήθησε πολλούς νέους, ειδικά αυτούς που ήθελαν να βοηθηθούν. Τώρα όμως θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς που είναι αδρανείς και Θέλουμε να αρχίσουμε από την αρχή του 2021 όταν θα ξεκινήσει η εφαρμογή των νέων μέτρων του Κοινωνικού Ταμείου για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσουμε να τους κινητοποιήσουμε. Δεν θέλουμε δηλαδή να περιμένουμε να γίνει το κακό σε μια περιφέρεια και μετά να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο. Ε, να μπορούμε δηλαδή έτσι να τους βοηθήσουμε δίνοντας ευκαιρίες της απασχόλησης ή νέας κατάρτισης. Προτείναμε απλοποίηση της διαδικασίας για την κινητοποίηση. Τώρα χρειάζεται να ληφθούν δύο αποφάσεις από τις δημοσιονομικές αρχές και πιστεύουμε πως αυτό δεν βοηθά στην ταχύτητα, αν και το Ταμείο Προσμιοποίησης ανέκαθεν έφερε τον τίτλο του μέσου επίγουσας ανάγκης, έκτακτης ανάγκης. Αλλά δεν το χρησιμοποιούμε πια αυτό γιατί μέχρι που να πάρουμε εμείς απόφαση έχει περάσει η επίγουσα ανάγκη. Ποσοστά συγχρηματοδότησης. Τα έχουμε ευθυγραμμίσει στο υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης στα κράτη. και δεν θέλαμε να υπάρχει, γιατί δεν θέλαμε να υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στο Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Για τα κράτη-μέλη όπου η συγχρηματοδότηση είναι χαμηλότερη, είναι ενδιαφέρον γιατί έτσι παίρνουν ψηλότερο προ... Ε, προπολογισμό, συγγνώμη, περισσότερα χρήματα. Έτσι θα είναι καλύτερο για τα άλλα κράτη να χρησιμοποιήσουν το κοινωνικό ταμείο και να μην ε, ασχοληθούν με την ανάπτυξη ενός ειδικού project. Εναρμονίζοντας ε, τα ποσοστά σε χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, πιστεύουμε πως θα κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη ώστε να χρησιμοποιήσουν περισσότερο το Ταμείο παγκοσμιοποίηση σε περιπτώσεις μαζικών απολύσεων. Προτείναμε επίσης τον κανονισμό υπάρξει το πλαίσιο συγκεκριμένης παρακολούθησης των επιδόσεων με συγκεκριμένους δείκτες. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν ήδη τμήμα θα έλεγα του σχήματος. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς έτσι ώστε όσοι προετοιμάζουν κάποια προγράμματα να γνωρίζει εκ των προτέρων τι ε, ενημέρωση θα πρέπει να κάνει σε σχέση με την πορεία Περιεργώς στο Συμβούλιο κάποια κράτη-μέλη διαφώνησαν γιατί τα κράτη-μέλη τα οποία είχαν τηρήσει αυτές τους κανόνες ε, είχαν αν θέλετε ε, προβλέψει και την δυνατότητα ε, παρακολούθησης ελέγχου αναφοράς όπως θέλετε. Κάναμε και μία ε, ε, στο διαδίκτυο έρευνα έτσι ώστε να συλλέξουμε τις διαφορετικές ε, εμπειρίες, έτσι ώστε να δούμε ακριβώς το EGF σε ποιο βαθμό βοηθά τους δείκτες απασχόλησης και σε ποιο βαθμό αυτοί οι οποίοι υποστηρίχθηκαν από το EGF έχουν βοηθηθεί στο να βρούνε ε, μία θέση απασχόλησης. Στη νέα πρόταση αυτό θα περιλαμβάνεται σαν απέτηση. Η κυρία Μπλίνκεβιτσι αναφέρθηκε στις προετοιμασίες των τριών θεσμικών οργάνων για τον κανονισμό ε, του Ταμείου μας. η Ολλανδία, η Σουηδία ήταν κατά ε, της πρότασης για τον κανονισμό, η Φιλανδία τήρησε στάση αποχής, αλλά με τον κανόνα της πλειοψηφίας ε, ε, ελπίζω ότι στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε, μια, σε ένα λειτουργικό κυρίως κανονισμό του συγκεκριμένου ταμείου. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο τον οποίο θέσατε στη διάθεσή μας. Οι σκιώδεις τώρα έχουν τον λόγο και μετά τα υπόλοιπα μέλη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια και ευχαριστώ τη συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι σε πάρα πολλά σημεία δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει όμως ένα θέμα, το θέμα της διεύρυνσης του Ταμείου αυτού, της εμβέλειας του Ταμείου αυτού. Καταρχάς εμείς θα εγκρίνουμε τον Brexit και το θέμα των μελλοντικών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάτι το οποίο παραμένει ανοιχτό και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να προσαρμοστούν στην κατάσταση μετά από την αποχώρηση του ΙΤΑΒ. Νομίζω ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να ε, συμφωνήσει στη διεύρυνση της εμβέλειας. Υπάρχει επίσης και το θέμα της μετάβασης στους τομείς της ψηφιοποίησης και ε, του κλίματος δεν περιλαμβάνονται ε, στην εμβέλεια ε, του ταμείου αυτού παρότι είναι σημαντικά φαινόμενα. Δεν μπορούμε από τη μία εμείς να λέμε πόσο σημαντική είναι αυτή η τομή και τους εργαζομένους να τους αγνοούμε στην πρότασή μας. Είναι λοιπόν βασικό να διευρυνθεί η εμβέλεια, το πεδίο δράσης ε, του συγκεκριμένου ταμείου. Τώρα σε σχέση με το, με επόμενο πολιετές δημοσιονομικό θα πρέπει να υπάρξουν οι σωστές προβλέψεις για την χρηματοδότηση του Ταμείου που μας ενδιαφέρει. Προσβλέπω λοιπόν συνάδελφοι ε, σε γρήγορα βήματα προόδου. Ε, αυτό είναι προς όφελος των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μπρόφη, ευχαριστώ συνάδελφοι. Χθες σε μία από τις τελικές συμμετοχές μου σε ψηφοφορίες υπεψήφισα το να ξεκινήσουν οργανικές διαπραγματεύσεις για το Ταμείο αυτό για την παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι αυτά γίνονται με βάση το κείμενο το οποίο ψηφίσαμε πέρυσι. Βέβαια όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις εγώ δεν θα είμαι πια σκιώδης. Εύχομαι σε όλους επιτυχής διαπραγματεύσεις. Ελπίζω ότι το τελικό κείμενο στο οποίο θα καταλήξετε θα είναι κάτι το ιδιαίτερα χρήσιμο. The Τελευταία κυρία Φίλιπς από πλευρά των Πρασίων που απουσιάζει η κυρία Βαν Σπάρεντακ. Η Αλεξάνδρα Φίλιπς είναι σκιώδης, αλλά και εκείνη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ λέγομαι Κιμ Βαν Σπάρεντακ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς οι πράσινοι αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη μετάβαση προς ε, βιώσιμες ε, κοινωνίες περιβαλλοντικά εδώ και χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της διαδικασία οι απολύωμενοι εργαζόμενοι ε, εταιριών σε ανασυγκρότηση και χρειάζεται υποστήριξη ε, ακριβώς αυτός ο κόσμος για να βρει ποιοτικέ και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Χαίρομαι εξ ονόματος της ομάδας μου που έχει συμπεριληφθεί και αυτή η κατηγορία, γιατί θα πληγούν από την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα ή στην ψηφιακή οικονομία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ξέρει αυτό, αλλά θα ήθελα να μας εξηγήσει ε, ποιες είναι οι πιθανές συνέργειες που βλέπει ανάμεσα στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Και όπως και η συνάδελφος, θα ήθελα λίγο να με ενημερώσετε περισσότερο για την υπόθεση Καρφούρ και τι συμβαίνει εκεί ακριβώς. Κανονικά θα ήταν η κυρία Λίτση από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία, οπότε θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, στην ε, κυρία Σίτλο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό για ένα ταμείο να έχουμε ε, πάντα υπόψη μας ότι οι λύσεις τις οποίες προσδοκούμε να είναι σωστές λύσεις και να φτάνουν στους πραγματικούς ε, δικαιούχους και εκείνους που έχουν ανάγκη τα χρήματα. Η ψηφιοποίηση είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Μας τα είπανε και οι εργαζόμενοι στο Καρφούρ αυτά γιατί λέει όλο και περισσότερο υποστηρίζεται η ε, διαδικασία αυτή του λιανικού εμπορίου από την ψηφιοποίηση, δηλαδή το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο κόσμος ε, πλέον ψωνίζει διαδικτυακά. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να αντέξουμε στις προκλήσεις. να βοηθήσουμε πραγματικά αυτούς. On behalf of Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Γουσμάου αποφασιάζει. Αυτή ήταν η ε, σκιώδης. Η κυρία Γιονκέριος έχει ζητήσει το λόγο και άλλη μια συνάδελφος. Παρακαλώ. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση γιατί έχουν αναφερθεί οι προλαλήσαντες. Με αυτή τη νέα θητεία μήπως θα μπορούσαμε ε, να ε, μάθουμε πώς θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τέτοιες περιπτώσεις τύπου Καρφούρ. Το Συμβούλιο αρνήθηκε ε, να στήριξει την επιχείρηση αυτή. Τώρα αυτό έχει τελειώσει, δηλαδή επειδή λέει όχι το Συμβούλιο υπάρχει καμιά δυνατότητα προσφυγής κάπου να καταφύγουμε ενδιαφέρομαι να μου πείτε τι έγινε με το Καρφούρα, αλλά ρώτησαν και άλλοι συνάδελφοι. Ε, κυρία Ρεντέν, ευχαριστώ κυρία Βετγέν. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους και εισηγητές για το εξαιρετικό τους έργο. Ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση. Ε, συμφωνούμε όλοι ότι αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι πραγματικό εργαλείο ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ε, για τους εργαζομένους που απολύονται. Και δεν χωρά καμία αφιβολία ότι είναι χρήσιμο πραγματικά. Χαίρομαι για τις προτάσεις που θυμήσατε. Ε, ήταν και προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σχετικά με το ε, αριθμό των εργαζομένων μιας εταιρείας για να έχει πρόσβαση σε αυτό το ταμείο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο η μεταβλητή προσαρμογή, η παγκοσμιοποίηση, είναι η ψηφιοποίηση, δυστυχώς το Brexit και λυπούμαστε γι' αυτό και κάποια άλλα. Και η μετάβαση προς μια ουδέτερη κλιματικά ε, οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά ε, την περασμένη εβδομάδα έκανε την πρότασή της για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στα πλαίσια της Νέας Πράσινης Συμφωνίας και θα ήθελα παρακαλώ να με ενημερώσετε ε, πώς θα συνδυαστεί το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Φυσικά δεν θα είναι πάντα παράλληλα και ε, μπορεί να έχουν χρονική διαφορά μεταξύ τους τα ταμεία, αλλά Πώς θα φροντίσετε να γίνει σωστά η εφαρμογή και με στρατηγικό τρόπο για να ε, βοηθούμε τους εργαζομένους και γενικά τους πολίτες στην Ευρώπη. Η κυρία Ραφάλσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Έχω μερικές ερωτήσεις κι εγώ η σημαντικότερη είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου. Η τροποποίηση των συντελεστών συγχρηματοδότησης κλπ. Εμείς θέλουμε να διευρύνουμε την πρόσβαση στο Ταμείο, αλλά δεν αυξάνεται η πρικοδότησή του ε, σημαντικά. Εντάξει, από 170 εκατομμύρια έχουν γίνει 230. Είναι μικρή αυτή η αύξηση και φοβάμαι ότι επειδή ακριβώς έχει διαβρεθεί το πεδίο εφαρμογής, ε, φοβάμαι ότι δεν θα φτάσουν τα κονδύλια αυτά. 150.000 ε, ε, είναι οι εργαζόμενοι που θέλουμε να υποστηρίξουμε, άλλες πολλές χιλιάδες οι νέοι, δεν αρκούν οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχω και άλλη ερώτηση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία και το Ταμείο Προσαρμογής Παγκοσμιοποίησης. Αυτά τα δύο πώς συμπεριφέρονται το ένα προς το άλλο. Γιατί υπάρχουν ε, κάποιοι φόβοι για την απασχόληση ε, στην ε, χαλιβουργία, στο κατασκευαστικό τομέα, στις εξορυκτικές επιχειρήσεις. εκατοντάδες χιλιάδες θα είναι εκείνοι που θα κινδυνεύσουν να χάσουν τη δουλειά τους. Αυτοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Δεν θα πρέπει να στηρίζουμε μόνο τους νέους, αλλά και εργαζομένους. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στην εισηγήτρια για να κλείσει η συζήτηση αυτή. Παρακαλώ να μιλάτε όλοι πιο αργά. Γιατί εδώ ανάβουν διάφορα φωτάκια, μου στέλνουν μηνύματα και δεν ξέρω. Όλοι να μιλάμε πιο αργά. Κυρία Σουκόβα. Ευχαριστώ. Προσπαθώ, αλλά ξεχνιέμαι. Σας ευχαριστώ για τις θέσεις τις οποίες εκφράσατε. Το θέμα είναι να συνδυάσουμε τα τρία αυτά επίπεδα ε, γύρω από τα θέματα της παγκοσμιοποίησης. Έτσι και αλλιώ τα δύο πρώτα προγραμματίζονται εξ αρχής της προγραμματικής περίοδου, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι πολίτες ε, για την δίκαιη μετάβαση, να βρουν μια πιο καλή θέση απασχόλησης ή θέση απασχόλησης απλά, και σε σχέση με το κοινωνικό ταμείο ΣΥΝ να υπάρξει ακόμα καλύτερη ε, βοήθεια και παροχή υπηρεσιών στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό εφαρμόζεται για όλους και προγραμματίζεται για την περίοδο 23-27. Τώρα για το Ταμείο Μετάβασης ε, είναι επενδυτικό ουσιαστικά σε, σε περιφέρειες όπου οι δυσκολίες για το πέρασμα στην παγκοσμιοπέμινη οικονομία είναι οι πιο δύσκολες. Είναι ε, περιοχές με υψηλές, ε, υψηλά επίπεδα παραγωγής λιγνίτη ε, και υψηλά επίπεδα παραγωγής αερίων του καυσαερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε οι συνέργειες ανάμεσα στο κοινωνικό πλάς και στο ταμείο αυτό και σε όλα τα άλλα μέσα να καταστούν αποτελεσματικές και να έχουμε καταλήξει πριν από την κατάθεση των προτάσεων για την επόμενη προγραμματική. Θα πρέπει να εντοπίσουμε τις περιοχές αυτές και τις χώρες οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν τις πιστώσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες. Μια άλλη διαφορά είναι ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης περιλαμβάνει εννέα διαφορετικά μέτρα τα οποία συμπίπτουν ε, με ε, κάποια χαρακτηριστικά ε, των επενδύσεων του Κοινωνικού Ταμείου και του Περιφερειακού Ταμείου, αλλά ταυτόχρονα θα είναι πολύ πιο στοχευμένα. Η σχεδίαση τώρα και ο καθορισμός των περιοχών αυτών θα ξεκινήσει με τις εκθέσεις αναχώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από το Φεβρουάριο και μετά. Θα προσαρτήσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα διευκρινίζει ε, ποιες είναι οι περιφέρειες με τις ε, μεγαλύτερες ή τις περισσότερες ε, δυνατότητες έτσι ώστε οι, οι παρεμβάσεις του Ταμείου να συμβαίνουν εκεί όπου χρειάζεται και να βοηθούν και τους εργαζομένους αλλά και τις μικρομεσαίες φυσικά να βοηθούν την έρευνα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής και ε, να βοηθηθούν αυτοί που χάνουν την απασχόληση, την θέση εργασίας τους ε, να ανακτούν περαιτέρω ικανότητες επαγγελματικές και γνώσεις. Το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση θα παρεμβαίνει μόνο όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μαζικές απολύσεις. Το κοινωνικό ταμείο και το περιφερειακό προσπαθούν να αποφύγουν αυτές τις απολύσεις. Προσπαθούν να βοηθήσουν ε, καθ' την μεταβατική περίοδο να αποκτήσουν νέες ικανότητες ε, ή να βρουν μια άλλη θέση απασχόλησης. ενώ το Ταμείο για την Δίκαιη Προσαρμογή είναι κάτι το οποίο ε, θα καλύψει τις ανάγκες αυτών που ήδη έχουν χάσει τις θέσεις τους. Α, αν υπάρξει και μάλιστα μία μη αναμενόμενη επίπτωση στις επιχειρήσεις ε, των περιοχών αυτών ή και κάποιων άλλων περιοχών, τότε οι επιχειρήσεις αυτές πολλές φορές αναγκάζονται να απολύσουν σημαντικά ασημαντικούς αριθμούς εργαζομένων, οπότε το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει την παρέμβαση του EGF. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα τοπικής αν θέλετε κινητοποίησης. Εμείς έχουμε ε, αναφερθεί στην ψηφιοποίηση, στην αυτοματοποίηση, είναι προκλήσεις για όλο τον κόσμο που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πάντες και εμείς κάνουμε κάποιες προτάσεις για την αλλαγή του τύπου της βοήθειας την οποία λαμβάνουν αυτοί που χάνουν τις θέσεις απασχόλησής τους και προτείνουμε επιπλέον μέτρα έτσι ώστε να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις ή να βελτιώσουν τις υπάρχουσες. Νομίζω ότι όλα αυτά τα μέτρα χρειάζονται για όλους όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους. Στα πλαίσια του ισχύοντος ε, ε, πολιετούς δημοσιονομικού ε, οι περιπτώσεις βοήθειας εφόσον δεν συμφωνήσουν οι αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές κλείνει. Ε, υπήρξε ας πούμε στα πλαίσια του Κορεπέρ μια επιστολή προς το Κοινοβούλιο ε, ε, για το κλείσιμο της υπόθεσης του Καρφούρ. Ετοιμαζόμαστε να ενημερώσουμε τις τοπικές αρχές και θέλουμε να υπάρξει μια τροποποίηση βέβαια όπως είπαμε για τη διεύρυνση του στόχου, των στόχων του Ταμείου Δίκαιης Μετάφασης. Και μπορεί όμως οι τοπικές αρχές του Βελγίου να καταθέσουν εκ νέου αίτηση με κάποιες διαφοροποιήσεις ε, διευκρινίζοντας ακριβώς ε, καλύτερα τα πράγματα. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους διεύρυνσης του στόχου. Τότε αν είχαμε ήδη διευρύνει την εμβέλεια του Ταμείου, η υπόθεση Καρφούρ δεν θα είχε ε, κλείσει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ ε, να κλείσετε τη συζήτηση κυρία Πλίνκεβιτσίουτε. Ευχαριστώ την κυρία Σούκοβα. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση, για την εξαιρετική συνεργασία. Ε, ως εισηγήτρια πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η πρόταση. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, χρησιμοποιείται σωστά αυτό το ταμείο. Από το 2006 το έχουμε και λειτουργεί ε, και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε υπέρ των εργαζομένων και υπέρ των απολυμένων. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ τους και όδες Θα συνεχιστεί η συνεργασία για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Τελειώσαμε ε, τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ακολουθούν συντονιστές. Παρακαλώ να παραμείνουν οι συντονιστές στην αίθουσα.